Παράγραφος 11. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ψήφι Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, ας το ελέγξουν καλύτερα όμως. Άρα ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της ε, παραγράφου 11, αρχικό κείμενο άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Ευχαριστώ. Παράγραφος 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης δεκτή παράγραφος 13. Παράγραφος 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφορία. Κατάσταση στην Ταϊλάνδη. Κοινό ψήφισμα 7 πολιτικών ομάδων. Έχουμε μία τροπολογία στο ε, εκτιμώντας έμμα. Την τροπολογία είναι υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Και επομένως τώρα περνάμε στην ψηφοφορία, ε, ονομαστική ψηφοφορία του συνόλου του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, όχι, όχι. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τώρα κλείνω την ψηφοφορία. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Επόμενη ψηφοφορία είναι το θέμα μαζικές εκτοπίσεις παιδιών στην Ιγυρία λόγω των επιθέσεων της Μπόκο Χαράμ. Κοινό ψήφισμα 7 ομάδων. Παράγραφος 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό. Ε, θεολογική σκέψη 1, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε σύνολο ψηφίσματος ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ερχόμαστε στην περίπτωση του Αλή Μοχάμετ Αλνίμερ, κοινή πρόταση ψηφίσματος 8 πολιτικών ομάδων. Παράγραφος 1, ε, αρχικό κείμενο, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα επίσης με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 7 αρχικό κείμενο. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πριν την ειδωλική αναφορά 11, έχουμε τροπολογία 1, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ήταν σαφές. Εγκρίθηκε. Παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ερχόμαστε τώρα στο σύνολο του ψήφου να τους ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επόμενο. Η ψήφιση εκθέσεω Ταγιάννη, του Πρόεδρου Ταγιάννη, υπηρεσίε πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Επιτροπή Οικονομικών, Οικονομική και Νομισματική πολιτική. Ψηφίζουμε το κείμενο συνολικά. Α, έχουμε τροπολογία 1 ε, της Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση Κομισιόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα ονομαστικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία. Νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, η περίπτωση τη Ισπανία. Ψηφίζουμε αρχικά την, παράγραφο, την τροπολογία 8, σε μετά ονομαστικά έρχεται για το πρώτο τμήμα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, ονομαστικά και αυτό, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο της παραγράφου 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Πρώτο τμήμα επαναλαμβάνω υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Καταπίπτει. Θέλετε να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα. Μάλιστα. Ελέγχουμε το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα παραγράφου 3. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα θα ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα τώρα. Ψήφι υπέρ του δεύτερου τμήματος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τώρα, τροπολογία 9 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4, αρχικό κείμενο, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12, ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε σε παράγραφο 7. Αρχικό κείμενο, ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα παράγραφος 9, ονομαστικά, Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. Ο, εντάξει, θα το ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ήταν αμφίροπτο αποτέλεσμα. Μετά την παράγραφο 12 έχουμε την τροπολογία 13, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 19, το αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστικά, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. Τρίτο τμήμα ονομαστικά και αυτό άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Παράγραφος 20 αρχικό κείμενο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική σκέψη α. Τροπολογία 4. Ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα, στην ατολική σκέψη Β έχουμε τροπολογία 5 ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το B, το αρχικό κείμενο, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Εκλογική σκέψη Β, B. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προπολογία 6 τώρα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. Στο F έχουμε τροπολογία 1. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το F, το αρχικό κείμενο. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το G. Τροπολογία 2 ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται επομένως ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της ετολικής σκέψης G. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το H έχουμε την απολογία 3 ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Μετά την εντολική σκέψη I έχουμε την τροπολογία 7 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Έμμα, μη αρχικό κείμενο, ονομαστικά, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Το σκέψη ένα νη. Ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. The next vote is... Επόμενη ψηφοφορία. για τη θανατική ποινή. Έξι ομάδε έχουν υποβάλει κοινή σχεδία ψηφίσματο. Παράγραφο 1 του αρχικού κείμενο. πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, με ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συνάδελφοι, παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σα. Α, μα συγγνώμη, ήταν ονομαστικά. Παράγραφος 4. Αρχικό κειμένο. Λάθος, δικό μου. Παράγραφος 4. Αρχικού κειμένου δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Σαφές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7, ονομαστική κλίση. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Ονομαστική κλίση. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Ονομαστικά έναρξη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Αρχικού κειμένου ονομαστικά έναρξη ψηφοφορίας. Και πέρας. Εγκρίνεται επίση. Παράγραφος 14. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Επίσης εγκρίνεται λογική σκέψη νη. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχε. Επίσης εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο. Επόμενο ψήφισμα. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της Ερυθράς Ηλίου. πέντε έτη μετά το δίχημα. Σχέδιο ψηφίσματο. Ψηφοφορία. Παράγραφος 2. Αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχε. Επίση εγκρίνεται. Παράγραφος 5 αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την παράγραφο 17 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα από το τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Να το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ. Για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Με ονομαστική κλίση έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Παραγραφός 4. Με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στην παράγραφο 21 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 23. Αρχικού κειμένου με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εδηλική σκέψη 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σκέψη 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική σκέψη ε, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, άποχες. Αυτό το παρακαλώ για την τροπολογία 1, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται και τώρα να ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος. Με ονομαστική κλίση έναρξη παρακαλώ της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η επόμενη ψηφοφορία για την ανανέωση του σχεδίου δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα των φίλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο τη αναπτυξιακή συνεργασία. Περνάμε λοιπόν στην παράγραφο 2 αρχικού κειμένου με προφορική τροπολογία τη κυρία Λίντα Μακέβεν. Έχετε το λόγο κύριε Μακάβεν. Πάνε, ναι, λειτουργεί το μικροφωνό μου. Μία προφορική τροπολογία, επειδή τώρα η Επιτροπή ε, δημοσίευσε πλέον το, σχέδιο, το έγγραφο εργασία ε, ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή το θέμα αυτό. Ουσιαστικά μία ενημέρωση. Υπάρχει αντίρρηση, λέει η Πρόεδρος, ένσταση. Δεν είσαστε 40 όμως, άρα θα ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο και θα ψηφίσουμε την παράγραφο όπως τροποποιήθηκε προφορικά, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 10. Το αρχικό κειμένο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές και αυτό εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Με ονομαστική κλίση έναρξη παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση έναρξη. Πέρας. και απορρίφθηκε. Καταπίπτει λοιπόν το δεύτερο τμήμα και περνάμε έτσι στην ψηφοφορία στην παράγραφο 19 αρχικό κείμενο δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Έτσι λογική σκέψη. Ε αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Παρακαλώ πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό έγκρινεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος, παρακαλώ. Έναρξη της ψηφοφορίας ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και περνάμε λοιπόν έτσι στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα, στην έκταση τη κυρία Αμπόρσκα σε ό,τι αφορά τι ίσε ευκαιρίε και την ίσια μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασία και απασχόληση. Πρώτα να ψηφίσουμε την παράγραφο 1 του αρχικού κειμένου, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχέ, Απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε για να είμαστε και σίγουροι, παρακαλώ. Δεύτερο τμήμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία έναρξη. Πέρας τώρα. Α, βλέπετε. Απορρίφθηκε με διαφορά μίας ψήφου. Συνάδελφοι, αυτά συμβαίνουν, ξέρετε, στα κοινοβούλια. Παραγραφός 8 του αρχικού κειμένου σε τρία τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Και αυτό εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα παρακαλώ. Ονομαστικά έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη παραγραφός 9 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά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 Τέταρτο τμήμα. Παρακαλώ, έναρξη πληροφορία. Πέρας. Και εγκρίθηκε λοιπόν. Επόμενη είναι η παράγραφος 12. Με ονομαστική κλίση έναρξη, παρακαλώ. Πέρασα. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 13, αρχικό κειμένο. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Έναρξη. Πέρας. Εκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστικά πάλι. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα. Ονομαστική κλίση έναρξη. Πέρασε. Και αυτό εγκρίθηκε. Επόμενο παράγραφος 14. Αρχικού κειμένου σε Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας ελέγξουμε παρακαλώ, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ, ηλεκτρονικά. I close the vote. Εγκρίθηκε. Επόμενο, Παράγραφο 15 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό εγκρίνεται. Παραγραφός 16 του αρχικού κειμένου σε πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστικά έναρξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα ε, με ονομαστική κλίση έναρξη. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Η... Έναρξη. Πέρας. Και αυτό εγκρίθηκε. Τέταρτο τμήμα. Έναρξη. Πέρας. Και αυτό εγκρίθηκε. Πέμπτο τμήμα, ονομαστικά παρακαλώ. Έναρξη. Πέρας. Και αυτό εγκρίθηκε. Επόμενο, παραγράφος 17. Αρχικού κειμένου στο τρίτο τμήμα, τα πρώτα τμήμα. Με ονομαστική κλίση, έναρξη παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση έναρξη. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα ονομαστικά έναρξη πληροφορίας. Πέρας. Και αυτό εγκρίθηκε. Επόμενη είναι η παράγραφο 18. Πρώτη, τραπολογία 1, με ονομαστική κλίση, παρακαλώ. Έναρξη πληροφορία. Πέρα. Ναι, και. Παραγραφός 20 του αρχικού του κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 22. Με ονομαστική κλίση έναρξη παρακαλώ. Πέρας. Εκκριθήκε. Παράγραφος 23 του αρχικού κειμένου σου τμήματα από το τμήμα υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 24 παράγραφος αρχικού κειμένου υπέρ, κατά, αποχές και αυτό εγκρίθηκε. Παράγραφος 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. 25 διορθώνει πρόεδρο. Ή 25 διορθώνει πρόεδρο, συγγνώμη, του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ υπέρ κατά, αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 αρχικού κειμένου υπέρ, κατά, αποχές και αυτό εγκρίνεται. Παράγραφος 27, τροπολογία 3, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Να ψηφίσουμε λοιπόν την παράγραφο 27 του αρχικού κειμένου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Παράγραφος 28 αρχικού κειμένου σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, και αυτό εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Θέλετε, ζητείτε έλεγχο. Μάλιστα. Έναρξη ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα τη 28. Πέρας ψηφοφορία, παρακαλώ. Απορρίφθηκε διορθωριακά όμως το αποτέλεσμα, άρα μια... καλά κάναμε και το ελέγξαμε. Τρίτο τμήμα με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Επόμενη είναι παράγραφος 29, τροπολογία 4, υπέρ. Κάτα. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 30 του αρχικού κειμένου σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κάτα. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό εγκρίνεται. Η παράγραφος 31 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε γιατί δεν ήταν σαφέ. Γιατί την παράγραφο 31, δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφο 34. αρχή κοκκιμένου, στο τμήμα, τμήματα, παρακαλώ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Αποχέ. Έγκρινεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παραγράφος 36 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Παρακαλώ, πρώτο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Και απορρίφθηκε. Παράγραφο 36. Δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. Ονομαστική κλίση. Ένα ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Επόμενη είναι η παράγραφος 37 αρχικού κειμένου σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση, ένα ψηφοφορίας παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Επόμενη είναι η παράγραφος 37, δεύτερο τμήμα παρακαλώ, με ονομαστική κλίση, έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα με ονομαστική κλίση, παρακαλώ, έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Επόμενη πρώτο τμήμα. Ένταξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφο 42. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Με ονομαστική κλήση. Ένταξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 43. Αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό εγκρίνεται. Παράγραφος 44 του αρχικού κειμένου, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 45 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα 45 παρακαλώ με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 46 του αρχικού κειμένου. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Παράγραφος 50 με ονομαστική α, κλίση. Ένα ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 52. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Ζητείτε έλεγχος παρακαλώ. Εντάξει, ας ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη πληροφορίας. Πέρας. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε λοιπόν και το αρχικό κείμενο της παραγράφου 52 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίθηκε έλεγχος, μάλιστα, για την παράγραφο 52, ας ελέγξουμε παρακαλώ, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. 53 παραγραφό. αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εκριθήκε. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 45, 55, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 56. Του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφορίας. Πέρας. Και εγκρίθηκε λοιπόν. Η 13, θα ήταν 13, υπέρ. Κατά. Αποχές. Το εγκρίθηκε. Αν τη λογική σκέψη, C, με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Έναξη ψηφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε. Το D. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίθηκε. Ετολογική σκέψη G με ονομαστική κλίση άνοιξη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Η H, Ήττα. στα τρίτη μόδα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Μάλιστα, ζητείτε έλεγχο για το δεύτερο τμήμα λοιπόν. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορίας για το δεύτερο τμήμα του συλλογικής σκέψης ΙΤΑ. H. Ah, I, Πέρας ψηφοφορίας. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές και αυτό εγκρίθηκε. Ε, τη λογική μας, συνάδελφοι. Ήταν σαφέ το αποτέλεσμα και στην προηγούμενη ήταν σαφέ το αποτέλεσμα. Σα παρακαλώ, συνάδελφοι, ήταν σαφέ και θα συνεχίσουμε με την τελογική σκέψη Εντάξει, εντάξει, λέει ο πρόεδρο. Αφού κάνετε φασαρία, κερδίζετε. Τρίτο τμήμα, παρακαλώ, ελέγχουμε το τρίτο τμήμα τη τελογική σκέψη ήταν... Πέρας ψηφορίας. Απορρίφθηκε. Πολύ λυπάμαι συνάδελφοι. Ε, καλώς και το ζητήσατε, τα κάνετε και το ζητήσατε. Και περνάμε λοιπόν στην L. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Εγκρίθηκε, συγγνώμη. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στο Q τώρα με ονομαστική κλίση ένα ψηφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. ΤΑΦ. Ονομαστική κλίση. Έναξη ψηφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. Επόμενη είναι η τελική σκέψη W. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στο σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Yeah. And I'll close the vote and it has been carried πέρας ε, της ψηφορίας και εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι για την συνεργασία σας ε, στις ψηφοφορίες και τώρα περνάμε στις εκφυολογήσεις της ψήφου. We do a short break until we start with the explanation of the votes. Thank you, colleagues. Ξεκινάμε σε λίγο τις εκλογές ψήφου.